Έχουμε έναν συστηματικό διάλογο με τον Αντιπρόεδρο Κάλας από τότε που ε, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είχαμε όμως μία περίπτωση όπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Επίτροπος ήρθε και μίλησε ενώπιον του συνόλου της Επιτροπής μας. Πρόκειται λοιπόν για την πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Θα θυμάστε ότι στα τέλη Μαρτίου εγκρίναμε το πρόγραμμα εργασίας για το 2010 και αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να ζητήσουμε από τον Επίτροπο να μας και τις βασικότερες πρωτοβουλίες νομοθετικές και μη νομοθετικές οι οποίες θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του έτους και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε και κάποιες ε, προτεραιότητες για το 2011. Ξέρω κύριε Επίτροπε ότι ε, τα μέλη της ε, Επιτροπής θέλουν να συμποβάλλουν και ερωτήσεις για διάφορα ζητήματα και για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, πώς μπορούμε να σταματήσουμε τα ηφαίστεια, τέτοια πράγματα. και ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι όπως και ο ίδιος ότι πιστεύουν ότι θα έπρεπε να μπορούσαμε κάπως να σταματάμε και τα ηφαίστεια όταν εκρήγνεται. Υπήρχαν άνθρωποι που μου τηλεφώνησαν στο γραφείο μου κατά τη διάρκεια της, της περίοδου της εφηστιακής τέφρας που μου είχαν ερωτήσει τι κάνω εγώ για να σταματήσω το ηφαίστειο. Σας δίνω τώρα το λόγο για 10-15 λεπτά και στη συνέχεια οι συντονιστές που έχουν φτάσει πια στην αίθουσα θα σας υποβάλουν κάποιες ερωτήσεις και θα κάνουν σχόλια. Κύριε Επίτροπε, Αντιπρόεδρε Κάλλας, έχετε τον λόγο και σας παρακαλώ πολύ ας είστε ποικείς με τον Επίτροπο Κάλλας γιατί δεν το γνωρίζετε εσείς αλλά το ξέρω εγώ έχει ξεχάσει τα γυαλιά του. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Εντάξει. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και που μπορώ και μιλώ ενώπιον ε, του συνόλου της ε, Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Είχα και στο παρελθόν την ευκαιρία να μιλήσω με τους ε, συντονιστές για κάποια καυτά ζητήματα που είχαν να κάνουν και με το ηφαίστειο. Αλλά χαίρομαι που είμαι σε θέση αυτή τη φορά να μιλήσω με το σύνολο των μελών της Επιτροπής Μεταφορών. Το πρόγραμμα εργασίας έχει κάποιες, περιέχει κάποιες βασικές πρωτοβουλίες. Πρόγραμμα εργασίας λοιπόν της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα εργασίας δίνει τα αρκετές νέες προτεραιότητες στον τομέα των μεταφορών και το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την πολιετή διάσταση που θα μας επιτρέψει να μιλήσουμε για το 2010 αλλά και για τα επερχόμενα έτη. Προκειμένου να έχουμε μια υφόρο βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να καταφέρουμε να καταρρύψουμε τα διάφορα εμπόδια τα οποία υπάρχουν μέχρι στιγμή. Θα πρέπει να ανοίξει περισσότερο η εσωτερική αγορά και θα πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές προκειμένου να καταρριφθούν οποιαδήποτε εμπόδια που υπάρχουν. Το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματο και έχουν ήδη αναλυφθεί διάφορε πρωτοβουλίε για την προστασία των πολιτών με την ενδυνάμωση τη ασφάλεια και των δικαιωμάτων των επιβατών. Θα ξεκινήσω με τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον των μεταφορών. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τη βίβλο αυτή το Σεπτέμβριο και ελπίζω ότι θα έχουμε ήδη την πρώτη εκδοχή τον Δεκέμβριο. Και το πιο σημαντικό βέβαια να πετύχουμε την απαραίτητη ποιότητα στο έγγραφο αυτό, δηλαδή την ποιότητα του περιεχομένου. Το έγγραφο αυτό θα αναφερθεί στο μέλλον, στο όραμά μα για το μέλλον των μεταφορών, καθώ επίση και στι υποδομέ για τι μεταφορέ σε επόμενε δεκαετίε. Θα αναφερθεί στην καλή λειτουργία τη εσωτερικής αγορά, στην άπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώ επίση και τι νέε καθαρέ μεταφορέ και τα ευφύ συστήματα μεταφορών. Επίση, θα προτείνουμε μία ενσωματωμένη, ολοκληρωμένη προσέγγιση για τι υποδομέ και ένα σύστημα χρηματοδότηση. Η έκθεση του κυρίου Γκρός για το 2009 για το μέλλον της, των μεταφορών θα ληφθεί σαφώς υπόψη στην κατάρτιση αυτής της λευκής βίβλου. Του χρόνου θα έχουμε επίσης και μια αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα για τις μεταφορές t και θα ληφθούν αυτά υπόψη για το νέο πολιετές ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο. Πρέπει επίσης να έχουμε το απαραίτητο χρονοδιάγραμμα για το προπολογισμό αυτό και θα πρέπει να κάνουμε τη σωστή ιεράρχηση επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων. Θα έχουμε ένα βασικό πυρήνα ε, διαδρόμων βασικών αξώνων και αυτό το βασικό δίκτυο θα πρέπει να περιλαμβάνει καινοτόμε πράσινε τεχνολογίε. Έχουμε την απαραίτητη μεθοδολογία για να σχεδιάσουμε το νέο αυτό δίκτυο μεταφορών που θα πρέπει να συζητήσουμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα κράτη-μέλη. Η πρώτη σημαντική συνάντηση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε τις 10 T-Days στη Σαραγκώσα. Η από την Ισπανική Προεδρία, όπου θα μιλήσουμε και για τη στρατηγική χρηματοδότηση των δικτύων αυτών. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον κοινοτικό προπολογισμό, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τον κατακαιρματισμό που υπάρχει στα χρηματοδοτικά μέσα. Πρέπει λοιπόν όλη η χρηματοδότηση για τι μεταφορέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάδει με του βασικού στόχου που έχουμε θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τι μεταφορέ. Πριν το καλοκαίρι θα αναθεωρήσουμε την πρώτη δέσμη μέτρων για, το, για τους σιδηροδρόμους. Η αναθεώρηση αυτή θα δώσει μεγαλύτερη σαφήνεια και θα οδηγήσει σε καλύτερη εφαρμογή της πρώτης αυτής δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Θα ληφθούν υπόψη νέες ε, αρχές ε, τελών, καθώς επίσης και νέες ε, μορφές καταπολέμησης της ε, ε, ηχορύπανσης, καθώς επίσης και άλλων εκκρεμών ζητημάτων. Επίσης, θα ανοίξει η αγορά περισσότερο για τους επιβάτες, θα γίνει ο παρέτος διαχωρισμός ανάμεσα στην συνδρομική αγορά επιβατών και τη συνδρομική αγορά για τα προϊόντα. Αυτό αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητές μας για το 2011 και το 2012. Και ξέρω ότι η Επιτροπή σας επεξεργάζεται ήδη ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους και θα λάβουμε προφανώς υπόψη μας το ψήφισμα σας αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο στο σχέδιο πρότασής μας. Στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς θα παρουσιάσουμε τον Ιούνιο του χρόνου ένα νέο πακέτο μέτρων για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των λειτουργιών των αεροδρομίων και την καλύτερη χρήση των ικανοτήτων των αεροδρομίων, των υποδομών τους. Θα προτείνουμε να αναθωρηθούν τα και θέλουμε επίσης νέα μέτρα για την καλύτερη αξιολόγηση της ε, ικανότητας χωρητικότητας των αεροδρομίων. Θέλουμε επίσης να βελτιώσουμε τα συνδρομικά δίκτυα τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα προϊόντα το 2011 και θέλουμε και καλύτερη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων. Επίσης, ασφάλεια των επιβατών. Αυτό είναι ένα ακόμα θέμα. Θα ασχοληθούμε περισσότερο με τους ε, σαρωτές ε, σώματος, την αποτελεσματικότητα των σαρωτών αυτών και θα δούμε επίσης και τα ε, πιο λεπτά ζητήματα της εμπιστευτικότητας των δεδομένων και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Στόχος μου είναι να καταλήξουμε σε κάποια σχέδια κανόνων στα πλαίσια της διαδικασίας της επιτροπολογίας και οι κανόνες αυτοί να πάρουν τη συνέχεια τη μορφή κοινοτική νομοθεσίας. Επίσης, πριν το καλοκαίρι θα σας παρουσιάσουμε μία νέα πρόταση για την οδική ασφάλεια μέχρι το 2020, δηλαδή στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα πρέπει να καταφέρουμε πάντα στα πλαίσια βέβαια της επικουρικότητας να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές που υστερούν στα επίπεδα ασφάλειας για την οδική μεταφορά. Θα δώσουμε κάποιες, κάποιους βασικούς προσανατολισμούς και θα δημιουργήσουμε ένα, πλέον ένα πλαίσιο συνεργασίας με τα κράτη-μέλη και ένα πλαίσιο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συνεχίσει με την ίδια προσέγγιση όπως το εφιστάμενο σχέδιο δράσης και να θέσει στόχους οδικής ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως είχαμε κάνει και στο παρελθόν και όπως είχαμε δει άλλωστε και με την έκθεση Gross. Θέλουμε να διευκολύνουμε επίσης και την πρόοδο για την ε, διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια. Επίσης θέλουμε να επεξεργαστούμε μία πρόταση για να καταφέρουμε να ελέγχουμε καλύτερα τα οχήματα τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα παρουσιάσουμε μέχρι το καλοκαίρι και ένα νέο νομοθετικό πακέτο για τις ε, θαλάσσιες ε, μεταφορές. Θα πρέπει να καταφέρουμε να κάνουμε το θαλάσσιο τομέα, το ναυτιλιακό τομέα πιο ελκυστικό και θα πρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε και τις διατάξεις του Διεθνούς ε, Οργανισμού Θαλασσίων Μεταφορών προκειμένου να κάνουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανταγωνιστική στον θαλάσσιο τομέα. Πριν το τέλος του έτους θα υποβάλω μια αναφορά για, την, τα δικαιώματα των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Ουσιαστικά θα θέλουμε να δούμε αν με την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία προασπίζομαστε σωστά τα δικαιώματα των επιβατών ή αν χρειάζεται να ληφθεί επιπλέον δράση και θα έχουμε ενδεχομένω νέε προτάσει μέχρι το τέλο του έτου. Τώρα για την τεχνολογία. Όπω γνωρίζετε, η τεχνολογία αποτελεί βασική προτεραιότητα. Ήδη από τον Μάρτιο του χρόνου θα έχουμε το e-mobility package, ένα πακέτο μέτρων για, την, για τις νέες αυτές τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών. Θα έχουμε τα ολοκληρωμένα συστήματα σιδηροδρομικών εισιτηρίων, η ολοκληρωμένη χρησιμοποίηση ταχογράφων και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε στο μέλλον και να καταφέρουμε να καινοτομήσουμε κιόλα. Όσον αφορά την έρευνα για τις μεταφορές, του χρόνου θα παρουσιάσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για την ε, τεχνολογία στις ε, μεταφορές. Θα εντοπίσουμε τα, τους καλύτερους τομείς για την έρευνα με ορίζοντα το 2000 50 και θα επικεντρώσουμε πλέον την έρευνα σε κοινοτικό επίπεδο σε συγκεκριμένου τομεί. Η φεστιακή τέφρα, όπω το γνωρίζετε, μα έκανε να αποκομίσουμε κάποια μαθήματα και μα οδήγησε στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων. Είχα τη δυνατότητα να μιλήσω για το ζήτημα αυτό μαζί σα και στην Ολομέλεια. Το ζήτημα προφανώς μας απασχόλησε πολύ και παρακολουθούμε ακόμα και τις τελευταίες εξελίξεις. Μόλις χθες πήγα στον ε, Ευρωπαϊκό, μάλλον πήγα στον Ευρωκοντρόλ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας των Αεροπορικών Μεταφορών. Αναφέρθηκα σε κάποιες ε, προτεραιότητες. Ο κατάλογος αυτός βέβαια δεν είναι διεξοδικός. Θα υπάρξουν και άλλες προτεραιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας μου κάθε φορά που προκύπτει μια νέα δυνατότητα περαιτέρω νομοθεσία θα προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό και πιο σφαιρικό τρόπο να τα αποκρίνομαι στην ανάγκη αυτή και ελπίζω ότι θα έχω πάντα την υποστήριξη και την καλή συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα προσπαθώ πάντα να δίνω στο δυνατό μεγαλύτερη ορατότητα στον τομέα αυτό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα τεχνικός, αλλά πέρα από την τεχνική του διάσταση θα πρέπει να καταφέρνουμε να δείχνουμε ότι συμβάλλουμε περισσότερο για την καλύτερη διαβίωση στην Ήπειρό μας. Δεν αναφέρθηκα στη διεθνή διάσταση, ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι τη της πολιτικής μας. Κάνουμε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε, με την Βραζιλία επίσης έχουμε έντονε επαφές και θα κινηθούμε και προς ε, άλλες κατευθύνσεις και στο μέλλον. Ξέρετε ότι ιδίω στα πλαίσια της ενέργειας κυκλοφορίας μας ενδιαφέρει να έχουμε επαφές με πάρα πολλές χώρες, τρίτες χώρες και θα πρέπει να ισχύουν παντού οι ίδιοι κανόνες. Αυτά είχα να σας πω, με στη θέση για ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Σύντομη εισαγωγή, αλλά μεστή. Θα ήθελα πρώτα να έχουμε ένα γύρο με τους συντονιστές. Με ερωταπαντήσεις και κατόπιν γύρω με βουλευτές. Παρακαλώ, όποιοι θέλουν να μιλήσουν να το δηλώσουν. Θα σας διαβάσω το ονόματα των εγγεγραμμένων. Mr. Mrs. Mr. De Pasquale, Mr. So anybody else wants Όποιος άλλος θέλει να μιλήσει, να το δηλώσει παρακαλώ. Um, Για να μπει στον κατάλογο. Έχω μία ώρα περίπου. Um, Οπότε, Ματιέ, πρώτος είσαι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τις ε, απόψεις σας. Το πρόγραμμά σας ε, είναι μια πλατιά βεντάλια για τους ε, επόμενους μήνες και για τα επόμενα χρόνια. Γιατί όλα αυτά που ανακοινώσατε εσείς πρέπει να έχουν τύχει σωστής προετοιμασίας έτσι ώστε να μπορούμε να τα βιώσουμε το 2010. Κατά τη δική μου λοιπόν άποψη υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι συνάρτηση της επικαιρότητα, από την άλλη όμως έχει σχέση και με την κατάσταση που επικρατεί τώρα στις μεταφορές, όπου ανεξάρτητα από τα προγράμματα που παρουσιάζετε εσείς αυτή τη στιγμή, θα θέλαμε να γνωρίζουμε σε ποια κατεύθυνση θα ε, οδηγηθούν οι προτάσεις σας. Ας πάρουμε τους σιδηρόδρομους. Και θέλω να θέσω πολύ απλά το εξής ερώτημα. Προτίθεστε να προτείνετε το άνοιγμα της αγοράς. Και η συζήτηση αυτή θα ξεκινήσει τώρα, σύντομα, ή θα αφήσετε το Κοινοβούλιο και κάποιες μελέτες να ανοίξουν το δρόμο. Αυτό ισχύει και για άλλους ε, τομείς όπου ε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το άνοιγμα της αγοράς. Και σας ερωτώ απλά και μόνο για να ξέρω πώς αντιμετωπίζετε εσείς το μέλλον. Ε, θεωρείτε ότι εδώ μπορεί να γίνει μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο έτσι ώστε να έχουμε μια, ένα σταδιακό άνοιγμα στις οδικές μεταφορές γιατί το καμποτάζ αυτή τη στιγμή ε, προσωρινά τουλάχιστον είναι περιορισμένο. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τις απόψεις σας. και όσον αφορά την ναυτιλία έχουμε ε, λοιπόν ε, ε, μια κατάσταση που πάμε ένα βήμα μπρο και δύο πίσω. Και τι θα γίνει. Τον φάκελο αυτό προτίθεστε να τον εξετάσετε. Εγώ θα έλεγα ότι σε τελική ανάλυση εδώ έχουμε να κάνουμε με τομείς όπου θα βιώσουμε πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές συζητήσεις. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, σε άλλους τομείς. Θα ήθελα να γνωρίζω, σε σχέση με το ηφαίστειο, έχει τεθεί το θέμα της αποζημίωσης και θα ήθελα επ' αυτού να έχω ε, σαφή απάντηση εκ μέρου σας. Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε. Θα ξεκινήσετε συζήτηση για να εξτάσετε το ενδεχόμενο των αποζημιώσεων. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή η συμφωνία με τις ΗΠΑ πού ακριβώς βρίσκεται, το 2010 θα υπάρξουν νέε εξελίξεις. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον αν ε, η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο γενικότερα είχαν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν εκ των προτέρων. Επίσης, ε, είπατε ότι θα προβείτε ε, σε αλλαγή και αναθεώρηση των σλότ, των χρονοθυρίδων. Αυτό τι επίσης μια ερώτηση που τίθεται πολύ συχνά. Στα μεγατράξ, εσείς τι λέτε από αυτόν. Πολύ συχνά μας ρωτούν για αυτά τα μεγάλα φορτηγά. Ε, πολλοί θεωρούν ότι αποτελούν ε, τον ανταγωνισμό των σιδηροδρόμων. Ε, θα θέλαμε να γνωρίζουμε την άποψη σας από αυτόν. Τέσσερα λεπτά θα δώσω στον κάθε συντονιστή. Ο επόμενο είναι ο κύριο Αλκαντράουι και στου ευρωβουλευτέ δύο λεπτά για να θέσουν τι ερωτήσει του. Ο κατάλογο έχει γίνει μακροσκελέστατο. Τέσσερα λεπτά, ο κύριο Αλκαντράουι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση που μα κάνατε. Έχω επίγνωση ότι πολλά πράγματα βρίσκονται στα σκαριά, πολλές προτάσεις, αλλά ως ομάδα είμαστε και εμείς ανυπόμονοι, όπως είπε και ο Ματιέ. Βέβαια και εμείς έχουμε πολύ έργο μπροστά μας και πολλά θέματα να επεξεργαστούμε. Για το θέμα του ηφαιστείου, πριν από λίγες εβδομάδες μιλήσατε για μια μονάδα συντονισμού που θα πρέπει να συγκροτηθεί για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδου έκτακτες καταστάσεις. Αλλά δεν κατάλαβα τι καθήκοντα θα έχει αυτή η μονάδα συντονισμού, Πώ θα λειτουργεί και σε τι καταστάσεις θα επεμβαίνει. Γιατί δεν έχουμε μόνο εκρήξη φεστίων. Τι άλλα καθήκοντα θα περιλαμβάνει αυτή η ομάδα. Και κάτι άλλο που είπε ο Μάτια. Αναφέρθηκαν πολλά στον τύπο για την αποζημίωση και την αντιστάθμιση που θα λάβουν οι αεροπορικές εταιρείε για να χορηγήσουν τις αποζημιώσεις. Μερικές εταιρείε, για παράδειγμα, ε, μιλούν για αναβολή της εφαρμογής του συστήματος ε, εκπομπών προκειμένου να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις αποζημιώσεις τους. Εμείς διαφωνούμε βέβαια. Εσείς τι γνώμη έχετε. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για τους ε, εργαζόμενους στις ε, μεταφορές. Υπάρχει διάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα περιληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Η πρόταση σχετική καταρρίφθηκε στην Επιτροπή Απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να αναζητήσει μια λύση. Γιατί ε, αν επιβεβαιωθεί αυτή η θέση στην Ολομέλεια της Επιτροπής Απασχόλησης, οι αυτοαπασχολούμενοι θα περιλαμβάνονται κανονικά στο πεδίο εφαρμογή, ενώ εμεί θέλουμε μία συμβαστική πρόταση. Η Ευρωβινιέτα είναι ένα άλλο θέμα. Το Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2009, έχει, είχε αποκρισταλώσει τη γνώμη του. Πάει ένας χρόνος, περιμένουμε πολλά από το Συμβούλιο και τη Βελγική Προεδρία για να προχωρήσει αυτό το θέμα και διαρωτώ με η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την πρόθεση να ασχοληθεί με το θέμα της Ευρωβινιέτας και να ασκήσει πιέσεις για να επιτευχθεί επιτέλους συμφωνία. Και τέλος, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι οι ευρωβουλευτές να ενημερώνονται εγκαίρως για διάφορα μέτρα. Για παράδειγμα, το Σεπτέμβριο εγκρίναμε το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα. Υπάρχει όμως ένα χρονοδιάγραμμα. Προβλέπεται το 2010 να ληφθούν κάποια μέτρα, να ιδρυθεί ένα παρατηρητήριο για την κινητικότητα, ανταλλαγή απόψεων για τη χρέωση και το καθεξής. Μην ξεχάσετε λοιπόν, μην παραμελήσετε και αυτό το θέμα και μην αμελείτε να ενημερώνετε τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξέλιξη της κατάστασης κυρία Μάισνερ για Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάλλας για όλα αυτά που είπατε. Ε, πολύ έθιξαν θέματα που ήθελα να πω και εγώ, καλύφτηκα. Αλλά έχω πέντε βασικούς τομείς ε, που θέλω να σας αναφέρω. Το ένα έχει σχέση με χρήματα που δεν διαθέτουμε, δηλαδή ε, την αναστολή των bottlenecks και μετά όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα για τις μεταφορές. Αυτό θα αισθηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Σαραγκώσα. Ε, και για τα δύο θέματα, τα bottlenecks και τα TEN ε, πρέπει κανείς να διαθέτει κάποια χρηματοδότηση. Πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Ερωτώ λοιπόν, εσείς έχετε κάποια ιδέα, βεβαίως ε, είναι δύσκολο αυτό, αλλά πώς μπορούμε να βρούμε νέα ε, εργαλεία χρηματοδότησης για αυτούς τους τομείς για να χρηματοδοτήσουμε αυτά που είναι απαραίτητα. Άλλο τομέα. κοινή αγορά. Ε, εκεί το βρήκα πάρα πολύ καλό. Ε, είπατε ήδη στην αρχή ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους σας είναι η ολοκλήρωση της κοινή αγοράς στον τομέα των μεταφορών. Και αναφερθήκατε στα integrated ticketing, ενιαία έκδοση ειδηρίων, πολύ σημαντικό αυτό για τους επιβάτες στην Ευρώπη. Τώρα με το ηφαίστειο, αν υπήρχε αυτή η ενιαία έκδοση θα μπορούσαν οι ε, επιβάτες να επιστρέψουν πιο εύκολα στα σπίτια τους. Ε, δεν άκουσα όμως συγκεκριμένα στοιχεία. Πότε θα υπάρξει πια αυτή η ενιαία έκδοση. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά ίσως μπορείτε να μας πείτε πώς το βλέπετε χρονικά. Κατόπιν, διατροπικότητα. Και αυτό είναι ένα θέμα που ε, δεν νομίζω ότι μπορείτε να το αντιμετωπίσετε μόνο σας. Ίσως μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Το τρίτο θέμα σύντομο μιλήσατε για την ανταλλαγή εμπειριών ε, όσον αφορά την ασφάλεια στους δρόμους και μιλήσατε για διασωνοριακή υποδομή για την οδική ασφάλεια. Ε, και υπάρχουν και άλλα δύο θέματα. Τον Ιούλιο του 2011, αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι θέλετε να δημιουργήσετε τις ε, κοινωνικές προϋποθέσεις για τους ε, εργαζόμενους ε, στην ναυτιλία. Θέλετε να κατεθέσετε ένα συγκεκριμένο πακέτο και πρέπει να πω χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όλοι όσοι ασχολούνται με την ναυτιλία περιμένουν επιτέλους αυτό το πακέτο που θα καταστήσει το επάγγελμα πιο ελκυστικό. Τελευταίο θέμα η ηφαιστειακή τέφρα. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι τα δικαιώματα των επιβατών σε αυτήν την έκρηξη του ηφαιστείου δεν έγιναν σεβαστά όσο θα έπρεπε. Βεβαίω και υπήρξε μια ιδιαίτερη κατάσταση, αλλά ερωτώ εσά, εσεί τι λέτε, διαφυλάχθηκαν τα δικαιώματα των επιβατών ή όχι. Και όσον αφορά την ηφαιστειακή τέφρα, επειδή υπάρχει μια ομάδα κρούση, έχετε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ε, για το μέχρι πότε θα συνεχίζει να εργάζεται αυτή η ομάδα κρούσης. Ίσως να το είπατε στην αρχή, αλλά εγώ ε, δεν το άκουσα. Αλλά ξέχασα κάτι. Ο νέος ευρωπαϊκός ουρανός. Και αυτό είναι ένα θέμα που νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον. Υπάρχει τώρα ένας ε, νέος συντονιστής ε, που θα αρχίσει να εργάζεται. Νομίζω λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε ή ευχόμεθα να έχουμε ταχύτατη πρόοδο στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μέσνερ. Σχεδόν εξαντλήσατε το τετράλεπτό σας. κυρία... Ο κύριος Κράμερ πρώτα και μετά κυρία Λιχτεμπέργκερ. Ε, και εγώ ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ε, εισήγησή σα. Όσον αφορά τα bottlenecks, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Μόνο που η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα από 20 δις μειώθηκαν σε 8 δι. Τώρα βέβαια υπάρχουν νέε προτεραιότητε, αλλά δεν διαγράφηκε κανένα πρόγραμμα. Και θέλω να σα πω με κάθε ειλικρινία, εάν παραμείνουν αυτά τα τέσσερα μεγάλα ε, προγράμματα και το τελευταίο που είναι ε, η σύνδεση με τη Μεσίνα, ε, αυτά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να ελοποιηθούν γιατί δεν θα υπάρχουν χρήματα για όλα τα άλλα που είναι απολύτω απαραίτητα. Θέλω λοιπόν να σα πω ότι σήμερα στου σιδηροδρόμου τη Ευρώπη υπάρχουν λιγότερε σιδηροδρομικέ ποιες ε, διασυνδέσεις με το πρώην ε, σιδρούν παραπέτασμα από ό,τι υπήρχαν πριν από 20 χρόνια. Αλλά πρέπει να το προωθήσουμε αυτό, αλλιώς πώς να ενωθεί η Ευρώπη άλλο θέμα. Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020 για το κλίμα. Μείωση κατά 20% των διεξιδίων του άνθρακα. Αλλά αν δεν αλλάξει και το θέμα των μεταφορών δεν θα πετύχετε αυτό το στόχο. Το θέμα δεν είναι να μας παρουσιάζεται εμβαλωματικά διάφορα μέτρα. Αν δεν αλλάξουν οι συνθήκες πλαίσιο και εάν ε, δεν εισαχθούν ε, οχήματα και μέσα μεταφορά φιλικά προ το περιβάλλον, δεν θα πετύχετε το στόχο σα. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ, Ποιε είναι οι συγκεκριμένε πρωτοβουλίε που προτίθεστε να αναλάβετε για να αλλάξετε τι συνθήκε πλαίσιο. Όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείε. Ευρωπαϊκό οργανισμό έδωσε τα στοιχεία και βάσει αυτών οι ευρωπαϊκέ εταιρείε, αεροπορικέ μεταφορέ παίρνουν από τον φορολογούμενο κάθε χρόνο 30 δι ευρώ. Αυτέ ε, και να μην έχουμε τέφρα παίρνουν 30 δι ευρώ. Άρα δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, θα πρέπει να υπάρξει μια ανακατονομία, αλλιώς θα μπορέσετε να πετύχετε τους στόχους σας. Μιλήσατε για speed limits, ε, όρια ταχύτητας ε, και για το ενόπνευμα, για την επικουρικότητα σε αυτά τα θέματα. Εδώ συζητάμε και λέμε ότι θα πρέπει για λόγους ασφαλείας ε, και το πρωί να ανάβουν τα φώτα τα αυτοκίνητα. Όμως λέμε επίσης ε, δεν μπορούμε να υπάρχουν όρια ταχύτητας, δεν μπορούν να υπάρχουν όρια στην κατανάλωση υνοπνεύματος. Όλα αυτά είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Και τελικά τι γίνεται με την επικουρικότητα. Θα μπορούσαμε να συζητάμε και για τα, τις ε, ε αστικές μεταφορές, αλλά δεν ασχοληθήκαμε με αυτές και δεν τα καταλαβαίνω. Στις ε, μεταφορέ, μεταφορές, στην έκθεση Gross, προβλέπεται μέχρι το 2020 μείωση κατά τα 20%. Ε, αυτό τεχνικά μόνοι σα δεν μπορείτε να το πετύχετε. Εάν για μια τετραμελή οικογένεια στην Ευρώπη είναι πιο φτηνό να πάει στη Μαγιόρκα από το να πάει με το σιδηρόδρομο 200 χιλιόμετρα, αυτό δεν μπορείτε να το αλλάξετε αν δεν αλλάξετε τακτική και θα το πράξετε. Λοιπόν, θα αλλάξετε τακτική. Ένα σιδηροδρομικό είπε ότι οι αγορέ είναι κλειστέ, δεν έχουμε ανοιχτή αγορά και γι' αυτό ερωτώ. Ολοκληρωμένοι σιδηρόδρομοι χωρίς ε, να ανοίξει αγορά, αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά μη ολοκληρωμένη σιδηρόδρομη χωρίς άνοιγμα της αγοράς, αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Τι θα κάνετε με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στις μεταφορές. Τα ακούσαμε σήμερα. Υπάρχουν μερικές χώρες που λένε δεν με ενδιαφέρουν, δεν με ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εγώ θα κλείσω τα σύνορά μου. Εσείς λοιπόν τι θα κάνετε και κυρίως πότε. Θα περιμένετε πάλι 8 χρόνια όπως έγινε με το πρώτο ε, πακέτο το σιδηρομικό μέχρι να υπάρξει μια επίπληξη ή προτίθεστε να δραστηριοποιηθείτε πάρα αυτά για να επιπλήξετε εσείς τις ε, χώρες που δηλώνουν κάτι τέτοιο γιατί μπροστά στον νόμο είμαστε όλοι ίσοι. Η κυρία Φώστερ είναι η τελευταία μιλήτρια αυτού του γύρου από τους μεταρρυθμιστές συντηρητικούς. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλώς ορίσατε κύριε Επιτροπέ. Έχω τρεις ε, σύντομες παρατηρήσεις. Καταρχήν αναφερθήκατε στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον ενδεχόμενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενθαρρύνει τους σιδηρόδρομους προκειμένου να διοργανωθεί ένα ψηφιακό σύστημα κρατήσεων στην Ευρώπη για να μπορούν οι επιβάτες ταξιδεύοντας από τη Φιλανδία στο Μιλάνο να αγοράσουν τα εισιτήριά τους ε, από την αρχή και να μην χρειάζεται σε κάθε χώρα να αγοράζουν ξεχωριστό εισιτήριο. Νομίζω ότι αυτό επιθυμούν οι επιβάτες, να έχουν τέτοια δυνατότητα. Το ξανασκέφτηκε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να έχετε σχόλια σχετικά. Δεύτερο θέμα, η φεστιακή τέφρα. Σωστά είπατε ότι η συζήτηση στο Στρασβούργο ήταν ενδιαφέρουσα και επαναλαμβάνουμε ότι χαιρόμαστε για την έγκαιρη ενημέρωση που μας έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πολλά θέματα που θίξαμε. Βέβαια, παρόλο που γνωρίζουμε ότι οι χρήστες ε, και οι εταιρείε ε, θα ουσιαστικά είχαν μία απώλεια 1,7 δις ευρώ από το θέμα αυτό, το θέμα είναι πώς θα υποστηριχθούν οι αερομεταφορείς και οι επιβάτες. Θα υπάρξει αντιστάθμιση για τις εταιρείες για να δοθεί αποζημίωση στις, στους επιβάτες, αλλά δεν μπορούμε να αποκαλέσουμε μια τέτοια ενίσχυση κρατική επιδότηση. Κάτι αντίστοιχο είχαμε και με το κλείσιμο των αεροδρομίων κατά την τρομοκρατική επίθεση της 11 ε, Σεπτεμβρίου. Βέβαια, εδώ ήταν διαφορετική κατάσταση. Πώς θα βοηθήσουν όμως τα κράτη-μέλη της αερομεταφορικές εταιρείε που πραγματικά είναι στριμωγμένες εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Τώρα, για το δικαίωμα αποζημίωσης. Φυσικά θέλουμε να μπορούν να αποζημιώνονται οι επιβάτες και να μεριμνούμε για την τύχη τους, αλλά ήταν πραγματικά ανωτέρα βία και το κόστος είναι αποτρεπτικό εδώ οι αερομεταφορεί θα πρέπει να πάρουν κάποια χρηματοοικονομική ενίσχυση, ή μια αντιστάθμιση εξαιτία των έκτακτων αυτών συνθήκων και τη ανωτέρα βία που προέκυψε από την ΤΕΦΡΑ. Μπορείτε να μα δώσετε κάποια στοιχεία. Σε κάτι άλλο που αναφερθήκατε, τα, τους ερωτές σώματος, την πρόταση που θα υποβάλλεται στα μέσα Ιουνίου. Ε, ήταν αρκετά επίμαχο το θέμα και το θέμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ίδιο από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Γιατί το αεροδρόμιο Skip Hall, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί μηχάνημα που είναι υψηλή τεχνολογία, δεν δημιουργεί προβλήματα, ενώ άλλα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν μηχανήματα και μάλιστα προβλέπουν υποχρεωτική εφαρμογή του που θα δημιουργήσουν προβλήματα. Δεν ξέρω αν μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα διεκπεριωθεί το θέμα, αλλά τουλάχιστον δώστε μας κάποιες ενδείξεις για, το που στέκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θα είχατε καλοσύνη να απαντήσετε σε αυτό το πρώτο γύρο ερωτήσεων από τις πολιτικές ομάδες. Τέσσερα λεπτά. Πολύ δύσκολο μέσα σε τέσσερα λεπτά. Δεν μπορώ να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα γιατί ορισμένα θέματα είναι λεπτομεριακά. Ευτυχώς βέβαια πολλοί έθεσαν τι ίδιες ερωτήσει. Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικό. Το σιδηροδρομικό πακέτο θα το λάβετε το Σεπτέμβριο. Και φυσικά είμαι υπέρ του ανοίγματο των αγορών. Καμποτάζ. Είπε και στην αρχή ότι θα προτείνουμε κατάργηση του καμποτάζ στις οδικές μεταφορές. Για την ηφαιστειακή δέφρα. Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν για το ηφαίστειο. Βέβαια τα ηφαίστεια είναι ανυπάκουα. Αυτό είναι στοιχείο της ζωής, είναι κανόνας της ζωής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να δαμάσει τη φύση. Παρόλο που πολύ θα ήθελε. Αυτό είναι τμήμα του κινδύνου που εμπεριέχεται στις αερομεταφορές. Πάντως ο συντονισμός λειτουργήσε, κυρίως μεταξύ της ΕΑΣΑ και του Eurocontrol αλλά μερικές φορές οι εθνικές ε, εταιρείες, οι εθνικές υπηρεσίες αεροπορίας θα πρέπει να έχουν πιο άμεση δράση και καλύτερο συντονισμό, αν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν για τις αποζημιώσεις. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στο κείμενό της τουλάχιστον ήταν απερίφραση. Εμείς δεν μιλήσαμε για αποζημίωση, γιατί αποζημίωση σημαίνει ότι κάποιος ε, ε, είναι υπέτειο για κάτι, ζήμιο σε κάποιον και πρέπει να πληρώσει. Αλλά το κλείσιμο του εναέριου χώρου για λόγους ασφάλειας υπάκουσε σε κανόνες που εθετήθηκαν από όλους τους ενδιαφερομένους, από κοινού. Βέβαια, μερικοί θεώρησαν ότι αυτοί οι κανόνες θα έπρεπε να ήταν πιο ελαστικοί. Δεν ήταν δική μου γνώμη, αλλά ήταν κοινή απόφαση γιατί υπήρχε κίνδυνο για τα αεροπλάνα. Και αν γινόταν ένα τύχημα, ποιο ήταν υπεύθυνο για ένα τέτοιο αεροπορικό δυστύχημα, αν δίναμε την άδεια για τι πτήσει. Ήταν ενωτέρα βία, έκτακτο περιστατικό. Και τέτοιοι κίνδυνοι συμβαίνουν. Γι' αυτό οι συνέπειε θα πρέπει να τι αναλάβουμε από κοινού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μιλά για αποζημιώσει. Ούτε και για κρατικέ ενισχύσει. Βέβαια, αν κάποια αεροπορική εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα, μπορεί να υποβάλει αίτημα για κρατική ενίσχυση. Και αυτό προβλέπεται από τους υφιστάμενους κανόνες. Ο συνάδελφος Χωακίν Αλμούνια πρότεινε να εξετάσει ελαστικότητα αυτό το ζήτημα αν υποβληθεί, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα για κρατική ενίσχυση από καμία εταιρεία. Για τον το λόγο. Η ζημία ανέρχεται σε 1,7 με 2 δις. Όταν όμως έχουμε ένα έγγραφο που ζητά συγκεκριμένη κρατική ενίσχυση, το θέμα είναι διαφορετικό. Θα πρέπει να αποδειχθεί το κόστος, το ύψος της ζημίας. Η κρατική ενίσχυση είναι δυνατή, αποζημίωση όχι. Γιατί η απόφαση λήφθη από κοινού για διακοπή των πτήσεων, γιατί κατά τη γνώμη των ε, όσων έλαβαν την απόφαση, η ασφάλεια είναι πρωταρχικό αγαθό. Τώρα, κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει θέμα αποζημίωσης για τις ε, εταιρείες. Τώρα για τα δικαιώματα των επιβατών θα πρέπει να ισχύσουν οι διατάξεις για τα δικαιώματα των επιβατών. Και υπάρχουν τρία σκέλη εδώ, ενημέρωση, μέρημνα και η εναλλακτική πτήση ή αποζημίωση. Αν υπάρχουν υπερβολικές καθυστερήσεις, τότε αποζημιώνει η αεροπορική εταιρεία. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο ούτε εδώ. Ήταν έκτακτες οι περιστάσεις που οδήγησαν όλα αυτά τα προβλήματα και την αναστάτωση. Βέβαια υπάρχει και μια φαιά ζώνη και στο μέλλον θα πρέπει να προσέξουμε. Πάντως οι πιο σοβαρές ε, αεροπορικές εταιρείες ακολούθησαν τους κανόνες και φρόντισαν για τους, ε, τους δεν τους εγκατέλειψαν στη μοίρα τους. Πάντως το φθινόπωρο υποσχεθήκαμε να υποβάλουμε τις προτάσεις για αναθεώρηση και θα αντιλήσουμε πολλά συμπεράσματα και διδάγματα από αυτό το πάθημα. Αυτά για το ηφαίστειο. Α, και μία ερώτηση αν ζητήθηκαν εξαιρέσει από το σύστημα εμπορίας εκπομπών ή άλλες ε, ε, εκπτώσεις ή εξαιρέσεις. Και εγώ στις ειδήσει το άκουσα, αλλά επίσημα δεν υπευλήθη έτοιμα για παρέκκληση από το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Και αν κάποιος ε, δίνει μάχη για τα συμφέροντά του, το μείζον ζήτημα σήμερα, όπως είπατε κι εσείς πολύ με τις παρατηρήσεις σας, είναι ότι προτείνονται ακριβέστεροι δείκτη, δείκτες για τα όρια. Και μάλιστα συνεργαζόμαστε και με κατασκευαστές κινητήρων για να έχουμε σαφέστερη βάση για το τι περιορισμοί χρειάζονται στην κάθε περίπτωση. Και οι αεροπορικές εταιρείες πολλές φορές έρχονται και ζητούν με εκνευρισμό να απελευθερωθούν οι πτήσεις, να τους δώσουμε το δικαίωμα πτήσεις. Εντάξει, να τους δώσουμε το δικαίωμα πτήσεις. Αν όμως συμβεί κάποιο ατύχημα, ποιος θα είναι ο υπεύθυνος. Η τέφρα είναι επικίνδυνη. Ήταν αναφυσβήτητο αυτό. Έγινε μία πτήση στον έφος της ηφαιστειακής τέφρας και είδε φωτογραφία πώς κατήντεσαν οι μηχανέ μετά από τέτοια πτήση. Τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν ήταν φανταστικό αυτό ο κίνδυνο. Αυτά για το ηφαίστειο. Τώρα, σιδηρόδρομοι, τέντη, διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και θέματα χρηματοδότηση. Το θέμα αυτό είναι γενικό. Υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης σε ορισμένε περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Με το συνάδελφο Ιωάννης Χάν προσπαθήσαμε να συντονιστούμε στα διάφορα κοινά προγράμματα περιφερειακής πολιτικής για να τηρήσουμε τους γενικούς στόχους στρατηγικής. Ο κύριος Χάν μάλιστα θα έρθει στη Σαραγώσα και θα συμμετέχει στη συνδιάσκεψη αυτή για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Είναι πολύ σημαντικό γιατί τα περιφερειακά κονδύλια είναι πολύ πιο δαψίλη από ότι τα κονδύλια για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Πάντως υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τη χρηματοδότηση, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν επαρκώς ή αποτελεσματικά μέχρι στιγμής. Και θα το εξετάσω αυτό το θέμα, θα δω γιατί δεν έγινε αποτελεσματική χρήση αυτών των κονδυλίων, γιατί η χρηματοδότηση είναι προτεραιότητα για μας. Θα πρέπει να βρεθούν κονδύλια. Πολλοί αναφέρθηκαν στο θέμα της διαλειτουργικότητας και της ενιαίας έκδοσης εισιτηρίου. Αυτό πραγματικά είναι ένα μάθημα που έχουμε μάθει και ήδη προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για τέτοια ενημέρωση, ώστε να είναι δυνατή η ενιαία έκδοση, όχι μόνο ε, να έχουμε διατροπικά εισιτήρια αλλά και διατροπικά ωράρια και χρονοδιαγράμματα. Όχι μόνο για τις πτήσεις αλλά και για, τα, για τους σιδηροδρόμους. Να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες ε, πληροφορικές και επικοινωνίες για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο. Και αν ένας απλός επιχειρηματίας θέλει να στείλει ένα εμπορευματοκιβώτη από το σημείο Α στο σημείο Β, τι πληροφορίες θα έχει, τι δρομολόγια να ακολουθήσει, ποιους άξονες να χρησιμοποιήσει. Και ο κύριος Κράμερ πολύ σωστά είπε ότι υπάρχουν στενοποί. Μερικά προγράμματα είναι τόσο μεγαλεπίβολα που είναι και χρονοβόρα στην εφαρμογή. Πάντως καλύτερη οργάνωση απαιτείται και η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας θα μας βοηθήσει. Ευρωβινιέτα. Η Ευρωβινιέτα είναι ένα θέμα που επεξεργαζόμαστε από κοινού με την Βελική Προεδρία. Έχει κολλήσει κάπου. Στα δικαιώματα των επιβατών, πολλά προγράμματα και πολλές λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τα όρια ταχύτητας τώρα και τα όρια ενοπνεύματος. Η... Στη Γερμανία δεν υπάρχει όρια ταχύτητας είναι ίσως Η μόνη χώρα που δεν έχει όρια ταχύτητα. Αν όμω κανεί οδηγεί στη Γερμανία, διαπιστώνει ότι υπάρχουν πινακίδες που περιορίζουν την ταχύτητα. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να έχουμε ένα πανευρωπαϊκό όριο ταχύτητα ή ένα πανευρωπαϊκό όριο υνοπνεύματος, γιατί είναι διαφορετικέ οι κουλτούρε. και σε ορισμένες χώρες ε, ε, μπορεί κανεί να εμπιστευτεί του πολίτε σε άλλε χώρε δεν του εμπιστεύεται τόσο. Υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις κατανάλωσης και πνεύματος. Τώρα, η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογραφεί στις 30 Ιουνίου με την Ισπανική Προεδρία. Αλλά μέχρι να επικυρωθεί θα περάσει πολύ καιρό. Και πολύ σημαντικό είναι να υπογραφούν και άλλες παρόμοιες συμφωνίες. Εντάξει κύριε Επιτροπέ, καλά τα πήγατε, μια χαρά. Τώρα έχουμε όπως είπα ένα μακροσκελέστατο κατάλογο με μέλη της Επιτροπής που θέλουν να μιλήσουν. Θα σας περιορίσω σε ένα δίλεπτο, αλλιώς δεν θα προλάβουν να μιλήσουν όλοι και δεν θα απαντηθούν και οι απορίες σας. Θα κάνω ό,τι μπορώ πάντως για να υπάρξει ισόρροπη εκπροσώπηση. Ο κύριος Καντζάν, για δύο λεπτά κύριε Καντζάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και σας ε, καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Άκουσα αυτά που μας είπατε και πράγματι το πρόγραμμά σας είναι πολύ φιλόδοξο. Εγώ πρέπει να πω, έχω κάποια δυσκολία ε, αυτή την εποχή να ε, εργαστώ, διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα επιχειρήματα τα οποία αφορούν ε, στη δική σας τη θέση και στο γεγονός ότι μιλάμε για το σιδηροδρομικό πακέτο, την αναθεώρηση των ε, διευρωπαϊκών δικτύων, ε, τις εμπορευματικές μεταφορές. Σήμερα το πρωί με την έκθεση Gross ε, ασχοληθήκαμε με τις βιώσιμες μεταφορές στο μέλλον και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον προγραμματισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από την άλλη πλευρά ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Λευκή Βίβλος, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές για τον προγραμματισμό έχουν ήδη εκπονηθεί, άρα δηλαδή κατά κάποιον τρόπο πρέπει να καταλήξουμε σε ένα προγραμματισμό, σε μια κατευθυντήρια γραμμή για την διαλειτουργικότητα. Όλα αυτά έχουν σχέση και με τα δικαιώματα των επιβατών. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για τα δικαιώματα των επιβατών στα λεωφορεία Πούλμαν και στα σκάφη. Μας είπατε ότι του χρόνου ε, θα υπάρξουν ε, θέματα που αφορούν το σύνολο ε, των μεταφορών και της διαλειτουργικότητα. Εγώ εκεί που θέλω να σταματήσω και να κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση είναι το εξή. Εσείς ήρθατε εδώ και μα μιλήσατε για ένα ταμείο το οποίο θα έχει ως στόχο να εξετάσει τις ε, οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν. Πρώτα πρέπει να γίνει αυτό και μετά να συσταθεί ένα ταμείο. Εδώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω η Ευρώπη πού πρέπει να οδηγήσει την οικονομία της και νομίζω αυτός ο τομέας είναι καθοριστική σημασία και θα θέλαμε να ξέρουμε πώς ακριβώς σκέφτεστε από αυτού. Επόμενη κυρία Σάντα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να ερωτήσω το εξής. Η Κομισιόν πότε προτίθεται να καταθέσει νέα πρόταση η οποία θα, είναι, ε, θα σχετίζεται με το, τις διασυνοριακές ε, μεταφορές. Επίσης, ε, πιστεύετε ότι κάτι πρέπει να κάνετε για τις υποδομές. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει ένα πιλωτικό πρόγραμμα έτσι ώστε να ε, συμπεριληφθούν οι αρμόδιοι που ασχολούνται με τις ε, οδικές μεταφορές αλλά και άλλοι οι οποίοι θα μπορούσαν να μας ε, βοηθήσουν έτσι ώστε να έχουμε συνειδητοποιήσει περί ακριβώς πρόκειται στις οδικές μεταφορές κατόπιν όσον αφορά τον προϋπολογισμό των μεταφορών εγώ νομίζω ότι στον τομέα αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα στόχο μιλάμε για τον προϋπολογισμό, αλλά πρέπει να καταλήξουμε καταρχήν σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Κατόπιν, όσον αφορά την διακυβέρνηση. Εκεί προτίθεστε να προβλέψετε ένα συγκεκριμένο μηχανισμό έτσι ώστε να μπορείτε να εκφράσετε τα εθνικά συμφέροντα. Νομίζω ότι εδώ ε, χρειαζόμαστε μία πρόταση από πλευρά τη ε, Κομισιόν που να μπορεί να στηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ε, για τι θαλάσσιες μεταφορέ, για τα λιμάνια, την επιμελητεία, τεχνολογίες. Ακούσαμε ότι εδώ έχετε κατά νου ένα πρόγραμμα, ε, μιλήσατε για τον νέο ευρωπαϊκό ουρανό. Έχουμε την εντύπωση ότι πολλά γίνονται, αλλά κανείς δεν το κόστος. Ε, κατόπιν, ε, δικαιώματα επιβατών. Εδώ έχουμε τον τομέα των πούλμαν λεωφορείων και από την άλλη τις θαλάσσιες μεταφορές. Μήπως θα πρέπει να υπάρχει κάποια ενοποίηση έτσι ώστε οι επιβάτες να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις αυτά που ήδη απαντήσατε. Αυτά που είπε η συνάδελφος σχετικά με την Ευρωβινιέτα είπατε ότι το θέμα αυτό θέλετε να το συζητήσετε με την Βελγική Προεδρία. Ε, πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί μία πλειοψηφία και τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους την Ευρωβινιέτα και πώς ένα άλλο θέμα, πώς θα έχουμε μετακίνηση του μοντέλου, του προτύπου αν τελικά δεν εργαστούμε συστηματικά για να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη στον τομέα. Ένα ειδικό θέμα που με απασχολεί είναι κατά πόσον θα λάβετε μέτρα έτσι ώστε επιτέλους και ευτυχώς έχουν εντάξει τελειώσει οι εκλογές στην Ιταλία για να μπορέσετε να ασχολείτε πάλι με το πρωτόκολλο για τις Άλπεις ε, και για τις μεταφορές. Τώρα γίνεται να προχωρήσουμε. Επιτέλους ε, έγιναν αυτές οι εκλογές ε, στο Βένετο. Αυτή η ιστορία τώρα διαρκεί 15 μέχρι 20 χρόνια. Ε, σιγά σιγά νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Δύο ευρωπαϊκά δίκτυα. Η δική μου συγκεκριμένη ερώτηση είναι η εξή. Θα υπάρξουν αλλαγές στον κατάλογο των προγραμμάτων ε, στον κατάλογο των 30 ή μήπως ε, θα υπάρξει κάποια, θα οριστούν κάποιες ε, προτεραιότητες με βάση τους συντονιστές. Νομίζω εγώ δεν εκπλήσωμαι για το ότι δεν υπάρχει περαιτέρω οικοδόμηση και αυτό εξηγείται και από του προπολογισμού των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη δεν γνωρίζουν κατά πόσον οι γειτονικέ χώρε θα κάνουν κάτι για να προχωρήσουν οι μεταφορέ. Τέλο, όσον αφορά τη συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων, ε, ο χρόνο οδήγηση και ο χρόνο εργασία, αυτό δεν το απαντήσετε. Μήπω έχετε την καλοσύνη να τοποθετηθείτε από αυτού. Ο κύριο Αντεγκράντες Πασκουάλ. Ε, señor presidente, un día aquí lo pasará Μια μέρα τα περνάτε καλά, μια μέρα πιο δύσκολα. Ευχαριστώ για τη φιλοδοξία σας. Γιατί ενώ με συμμερούμε τώρα τελευταία για τις κρίσεις, είναι πολύ ελπιδοφόρο να βλέπουμε ένα τόσο μακροσκελή κατάλογο με μεγαλεπίβολα σχέδια. Γιατί είναι τόσο πλούσιο αυτό το μενού που μας παρουσιάζεται, πολύ φοβόμαι ότι δεν θα έχουμε ούτε χρόνο, ούτε κονδύλια για να το διεκπαιρεώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ευπρόσδεκτο το φιλόδοξο πρόγραμμά σα. Τώρα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Τι γίνεται με την κρίση που τα ταμείων είναι μείον και τα κράτη-μέλη είναι απρόθυμα να συμβάλλουν. Πώς θα διαλέξουμε τις προτεραιότητες για το ηφαίστειο. Έχετε δίκιο, δεν προσπαθούμε να ρίξουμε ευθύνη σε κανέναν, αλλά θα πρέπει να δούμε τι διδάγματα θα αντλήσουμε. Μήπως ε, εφόσον οι ασφάλειες καλύπτουν θεομηνίες, δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα ταμείο ειδικό για να αποζημιώσει τους επιβάτες για το σιδηρόδρομο. Πώς θα τελειώσει αυτό το όνειρο των νεόπλουτων για τα τρένα υψηλής ταχύτητας και για να βελτιωθεί η μεταφορά εμπορευμάτων μέσω των σιδηροδρόμων. Πότε θα ε, υλοποιήσουμε επιτέλους την απελευθέρωση και των λιμανιών, γιατί είναι ένα ένας παλιός πονοκέφαλος. Πιστεύω θα πρέπει να δείξουμε τόλμη και να περάσουμε στις πράξεις, να μην παραμείνουν στα λόγια αυτές οι προθέσεις. Επίσης, σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας για τα μέτρα βελτίωσης ασφάλειας στις οδικές μεταφορές. Ο κύριος Βαντάλεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι για τον πολύ φιλόδοξο κατάλογο των σχεδίων σας και των προτάσεών σας, αλλά λείπει ένα πολύ σημαντικό σημείο, μια έκθεση που συζητήσαμε εδώ και θα εγκριθεί στην Ολομέλεια. Πρόκειται για, τη, για τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις χώρες και για το πώς κοστολογούνται ουσιαστικά οι παραβιάσεις εμείς οι παραβάσεις. Θέλουμε μια ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων της οδηγίας ε, για το χρόνο οδήγησης και χρόνο ανάπαυλας. Πώς θα συμβάλετε, πώς θα επέμβετε, ώστε οι οδηγοί να μην πλήττονται από τις διαφορετικές διατάξεις που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Στην ε, εσωτερική αγορά πολλές φορές ε, συναντούμε μερικά παράδοξα παραδείγματα. Τα φίλτρα, για παράδειγμα, των αιωρούμενων σωματιδίων. Κάποιος ήθελε να αγοράσει ένα τέτοιο φίλτρο στη Γερμανία, αλλά δεν μπόρεσε γιατί ο Δανός ε, μεταφορές που ήθελε να αγοράσει το φίλτρο στην Γερμανία δεν μπόρεσε να το χρησιμοποιήσει στη Δανία, γιατί στη Δανία δεν αναγνωρίζεται, αναγνωρίζεται μόνο στη Γερμανία αυτό το φίλτρο. Πραγματικά υπάρχουν αλλοπρόσελες καταστάσει που δημιουργούνται στην εσωτερική αγορά. Χαίρομαι για την πρότασή σα για το καμποτάζ και για την πρόταση κατάργηση κυρίω γιατί το καμποτάζ δημιουργεί περιορισμό στην εσωτερική αγορά. Και για τα φορτηγά, όσο μεγαλύτερη είναι η τόσο το καλύτερο και για την αγορά και για το περιβάλλον. κυρία Τσικάου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το πρώτο μου ερώτημα έχει να κάνει με τους χρηματοοικονομικούς πόρους για την ε, περχόμενη περίοδο. Θα ήθελα να αφαιρθώ στον τρόπο με τον οποίο εσείς πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να βελτιώσετε και να αναπτύξετε περισσότερο τις μεταφορικές υποδομές στην Ανατολική Ευρώπη και επίσης πώς θα καταφέρετε να υποστηρίξετε τα ευφυή e συστήματα μεταφορών και πώς θα εγγυηθείτε την διαλειτουργικότητα των ε, συστημάτων αυτών. Πώς επίσης θα καταφέρετε να έχετε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ευρώπη. Από ό,τι φαίνεται θέλετε να δημιουργήσετε μια τέτοια στρατηγική για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές επίσης και θέλετε να λάβετε υπόψη σας διάφορες διαστάσεις, το περιβάλλον, τον τουρισμό, τους υφιστάμενους ε, λιμένες, ε, τη χρησιμοποίηση καυσίμων. Να καταγράψετε επίσης τους τόλους στο σύστημα πιστοποίησης και στο σύστημα εκπομπών. Θα ήθελα λοιπόν να μας στείλετε το γραπτό κείμενο βάσει του οποίου θα καταρτήσει το σύστημα αυτό για να είμαστε και εμείς σε θέση να επιτηρήσουμε την εφαρμογή του. Πρόεδρος, μπορείτε κύριε Επίτροπε σε 10 λεπτά να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις. Η τελευταία ερώτηση δεν είχε να κάνει με το πρόγραμμα εργασία. Το πρόγραμμα εργασία είναι επίσημο κείμενο το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σα έχει ήδη διανεμηθεί. Μπορείτε λοιπόν να παρακολουθήσετε εκ του σύνεγγυ στην εφαρμογή του. Όπω σα είπα, ενδεχομένω να προσθέσουν και κάποιε νέε ιδέε σε αυτό το πρόγραμμα εργασία. Πάντω σα έχει σταλεί. Τώρα, οι αυτοαπασχολούμενοι και τα μεγάλα φορτηγά, τα mega trucks Για τα τελευταία δεν μπορώ να σας δώσω σήμερα μία απάντηση. Αναφέρομαι στα μεγάλα επιμήκια αυτά φορτηγά τα οποία ονομάζουμε Megatrax. Ξέρετε, το βασικό ζήτημα όμως έχει να κάνει με το μήκος των οχημάτων αυτών. Πολλές φορές το μήκος τους αντιστοιχεί στο μήκος λεωφορείων τα οποία διασχίζουν ε, πόλεις. Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν τα φορτηγά αυτά, αλλά θέτουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Δεν υπάρχει παγιωμένη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμα για τα οχήματα αυτά. Επομένως υφίστανται ή τα πρότυπα τα οποία ήδη ισχύουν. δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο καθεστώ και έχει δοθεί πράσινο φω συγκεκριμένα για τα οχήματα αυτά. Όσον αφορά τώρα τα χρήματα και πόσα χρήματα θα ζητήσω, ξέρετε ότι ο προπολογισμό είναι κάτι το περιορισμένο ουσιαστικά. Το ξέρετε κι εσεί, είστε αρμόδιοι επί του προπολογισμού αρχή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάτε τις α, διάφορες προτεραιότητες για τον προπολογισμό και ξέρω ότι υπάρχει και έντονη διαμάχη πολλές φορές για το ποια προτεραιότητα είναι πιο σημαντική. Κυρία Αγιάλα, σαφώς θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα χρήματα στα πλαίσια του προπολογισμού, αλλά Ξέρετε κι εσείς πώς καταρτίζεται ο προπολογισμός. Δεν είναι εύκολο να ζητήσει κανείς το ένα δισεκατομμύριο ετησίως για τα τέντη t τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, μπορεί να δώσει όθηση αν μη τι άλλο σε κάποια project, σε κάποια σχέδια, αλλά πρόκειται για ένα ποσό το οποίο δεν αρκεί για να καλύψει όλα τα σχέδια. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στον κοινοτικό προπολογισμό, αλλά και τον προπολογισμό από τα κράτη-μέλη, από τράπεζες, από περιφέρειες, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι αυτοί μπορούν να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των ε, σχεδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πριν από λίγο καιρό ήμουνα σε, ένα, σε μια διεθνή συνδιάσκεψη για τις μεταφορές και θίξαμε ακριβώς και το ζήτημα αυτό, το πώς μπορεί να συμβάλλει και ο ιδιωτικός τομέας και πώς μπορούμε να έχουμε διάφορες περιπτώσεις συγχρηματοδότησης στις μεταφορές, τώρα για τους αυτοαπασχολούμενους. Η θέση μου είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν ε, έχω καμία πρόθεση να αναθεωρήσω την ε, θέση αυτή. Θα δούμε όμως αν, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν θα καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Ό,τι έχει προταθεί μέχρι στιγμής δεν αποτελεί συμβιβασμό. Πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική γραμμή. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσει ότι αυτοπασχολούμενοι θα πρέπει να ενταχθούν, τότε ναι, αυτό μπορούμε να το ακολουθήσουμε σαν εναλλακτική. Ενδεχομένως όμως να πει ότι θα πρέπει να μείνουν εκτός. Μέχρι στιγμή πάντω εγώ δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προ την πρότασή μα. Όσον αφορά τώρα την διασυνοριακή διάσταση, και κυρίως τα διασυνοριακά πρόστιμα. Ξέρετε ότι υπάρχουν διαφορετικές χώρες με διαφορετικά συστήματα επιβολής προστήμων. Έχουν ακουστεί διάφορες ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να εναρμονίσουμε τα συστήματα αυτά, πώς θα μπορούσαμε αν μη τι άλλο να αξιολογήσουμε καλύτερα τις πρακτικές, πώς θα μπορούσαμε να εναρμονίσουμε τις πρακτικές αυτές. Για τα διασυνοριακά πρόστιμα πάντως θα κάνω ό,τι περνάει από τα χέρια μου προκειμένου να επιλύσουμε το ζήτημα αυτό. Ξέρω το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα. Και βλέπετε ότι καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου στις Βρυξέλλες ε, έχουμε πολλά οχήματα που έρχονται από άλλες χώρες, ε, επιβάλλονται στα οχήματα αυτά πρόστιμα και βέβαια τα πρόστιμα αυτά δεν συνάδουν απαραίτητα με τα πρόστιμα τα οποία τα οχήματα αυτά θα είχαν δεχθεί αν κινιόντουσαν στην χώρα τους, στη χώρα προέλευσης. Πρέπει λοιπόν να επιληθεί το ζήτημα αυτό. Έχουμε επίση και το σιδηροδρομικό πακέτο, ζήτημα πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να γνωρίζω ακριβώ ποια κατάληξη θα έχει. Η Ευρωβινιέτα είναι επίση κέριο ζήτημα. Συμφωνώ και εγώ ότι. Ε, ενδεχομένω. Ε, να υπάρχει πρόβλημα στην προσπάθειά μας να φέρουμε σε εσωτερικό επίπεδο το εξωτερικό κόστος των, της, Ευρω, της Ευρωβινιέτας. Θα ζητήσω πάντως από τους αρμόδιους και τον προπολογισμό να μου πούνε αν είναι σε θέση να δώσουν τα απαραίτητα χρήματα και θα μπορούσαν να συμβάλλουν τουλάχιστον ορισμένες χώρες για το ζήτημα αυτό της ε, Ευρωβινιέτας. Έχω έρθει σε επαφή με διάφορες χώρες και βλέπω ότι αρχίζουν και συγκλίνουν πλέον κάπως οι απόψεις. Το σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μία χρηματοδοτική συνδρομή από διάφορες χώρες ε, μια συνδρομή η οποία θα μπορούσε να πάει προ ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο για τι Μεταφορέ. Ενδεχομένω από ένα Ταμείο Λιλεγγύη να μπορούσαν να έρθουν τα χρήματα αυτά. Για το ΣΕΖΑΡ τώρα. Δεν είπα αμφισβήτηση καθόλου. Το σχέδιο αυτό προχωράει όπω είχε προβλεφθεί στην αρχή. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί μετά το 2013. Πάντω είναι ένα πολλά υποσχόμενο σχέδιο και δεν νομίζω θα συναντήσουμε σημαντικά προβλήματα. Επομένω, θα διατηρηθεί ω έχει. Τώρα, οι σαρωτές ασφαλείας θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται και για τους λιμένες θα σας παρουσιάσουμε μία στρατηγική στα πλαίσια της οποίας θα θελήσουμε να θίξουμε και το ζήτημα της κατάρριψης των εμποδίων και της παροχής καλύτερων υπηρεσιών. Σας ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε. Τελευταίος γύρος ερωτήσεων. Ο κύριος Κόχ έχει το λόγο πρώτος. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Πέρα από τους long ε, εγώ Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια οδηγία έτσι και αλλιώ για το βάρος των ε, μεγάλων ε, φορτηγών. Δεύτερο ερώτημα. Νομίζω ότι οι πολίτες μας νιώθουν ασφαλείς γιατί ε, βλέπουν όλο και νέες διατάξεις από τις Βρυξέλλες. Αυτά που ήδη υπάρχουν πιστεύετε ότι μπορούν να ελεγχθούν, να προχωρήσουν και μάλιστα με αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φλάνκενστάιν. Κύριε Επίτροπε, τρεις ε, σύντομες παρατηρήσεις. Αφενός ε, θα ήθελα να επαναφέρω ε, την ερώτηση του κυρίου Γκρός αλλά να τη διατυπώσω με κάποιο άλλο τρόπο. Πιστεύετε κι εσείς ότι μπορεί κανείς να μάθει από τα λάθη του και ω εκ τούτου ένα port package 3 δεν τίθεται επιτάπητος. Επίσης είπατε ότι όσον αφορά το κοινωνικό ναυτιλιακό πακέτο. Κάτι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά ξέρετε, δεν πρόκειται μόνο για την εκπαίδευση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός αυτής. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον φορέα ΕΜΣΑ που εξετάζει το όλο θέμα και υποβάλλει τις σχετικές εκθέσεις. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη οποτεδήποτε καταρτίζει μια έκθεση. Το τρίτο που θέλω να πω, το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι μια δική μου παράκληση. Αποφασίσαμε να παρακαλέσουμε την Κομισιόν όσον αφορά ε, την ε, παρακολούθηση του διοξιδίου του άνθρακα το παρατηρητήριο αν θέλετε να κάνει κάποιες ε, εκτιμήσεις, κάποιες προβλέψεις και θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να έχουμε το στιγμό των δυνατών στοιχεία επ' αυτού. Ο κύριος Μπραντμπον, ε, δύο λεπτά. επιτέλους μου δώσετε και εμένα το λόγο. Ε, ένα θέμα σχετικά με την ηφαιστειακή τέφρα που το έθιξαν πολλοί συνάδελφοι. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι η Κομισιόν βεβαίω δεν μπορεί να κάνει κάτι για να εξαφανίσει αυτή την ε, τέφρα αλλά μπορεί να ρυθμίσει τα περί αυτής ε, γιατί ρυθμίζει τόσο άλλα και κάτι άλλο Μήπως έχετε ακούσει ποτέ ε, αυτό το πρόγραμμα που υπήρχε στη Βρετανική τηλεόραση, το περίφημο Yes Minister. Να σας πω γιατί το λέω. Γιατί εδώ έχω μία απάντηση σε μία κοινοβουλευτική ερώτηση, απάντηση από τον Επιτροπό ε, που δικαιώνει τον Sir Humphrey στο πρόγραμμα Yes Minister. Εγώ είχα θέσει μια πολύ απλή ερώτηση και η απάντηση είναι ε, μετά από τις διαμαρτυρίες που είχα λάβει από ε, ψηφοφόρους ε, μου ελέγχθη ότι ε, θα λυθεί το θέμα με τον κανονισμό που είναι γνωστός ως ΣΥΡΑ. Επειδή εδώ δεν πρόκειται για εμπορικές δραστηριότητες αλλά για χόμπι, εγώ είχα ερωτήσει κατά πόσον αυτά τα χόμπι θα μπορούσαν να εξαιρούνται από τον κανονισμό τη στιγμή που προσθέτουν ένα τεράστιο κόστος σε όσους ασχολούνται με τα χόμπι. Είναι δηλαδή δαπανηρά για αυτούς. Κοιτάξτε, εγώ Είμαι εδώ 11 χρόνια και αυτή είναι η χειρότερη απάντηση σε αυτά τα 11 χρόνια σε ερώτηση ε, που ε, υπέβαλα ποτέ. Δεν λέει τίποτα, ε, αχρηστή απάντηση και ερωτώ τον Επίτροπο τώρα. Κοιτάξτε, εσείς θα θελήσετε να δώσετε αυτή την εξαίρεση για όσους ασχολούνται με το άθλημα των πτήσεων εραστεχνικά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τα δίκτυα και τη χρηματοδότηση των δικτύων των διευρωπαϊκών και τις μεταφορές. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα νέο προσανατολισμό στη διακυβέρνηση και στη χρηματοδότηση των δικτύων αυτών. Έχετε αποφασίσει να κάνετε κατά μέτωπο επίθεση στα κράτη-μέλη εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε κι εσείς τους άλλους συναδέλφους Επιτρόπου σε άλλους τομείς για τα δίκτυα αυτά. Δεύτερο ερώτημα. Τι προτίθεστε να κάνετε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μη εφαρμογή της πρώτης δέσμης της ιδεοδρομικής από ορισμένα κράτη-μέλη ή αναθεώρηση του πρώτου αυτού πακέτου που ανακοινώνεται είναι ένας τρόπος να δημιουργήσετε εξαίρεση για τα κράτη-μέλη βάζοντας πάλι τον μετρητή στο μηδέν και δίνοντάς ουσιαστικά περισσότερο χρόνο για να συμμορφωθούν. Και τρίτη ερώτηση, όσον αφορά τους οργανισμούς. Ο... Οι οργανισμοί πλέον, οι υπηρεσίες, γίνονται ο ποδιοπομπαίος τράγος για πάρα πολλές πολιτικές Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτίθεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες αυτές στο όφελος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ανησυχώ πάρα πολύ για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών αυτών. Για παράδειγμα, η υπηρεσία για την χημική ασφάλεια κοστίζει πολύ περισσότερο, δέκα φορές περισσότερο από ότι η αρμόδια υπηρεσία για τις μεταφορές. Η ε, υπηρεσία για την συνδρομική ασφάλεια με τα χρήματα που έχει αποκλείεται να καταφέρει να επιτελέσει το έργο της και σε καμία περίπτωση θα επιτελέσει το έργο που πρέπει να κάνει για την ασφάλεια, την πιστοποίηση και τη λειτουργικότητα. ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ε, θα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τις ε, μεταφορές. Μιλήσατε για την κατάργηση των bottlenecks και ένα πρόβλημα είναι οι ε, μακροχρόνιες αυτές δικές και με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υπάρξουν έργα στον τομέα των μεταφορών. Χάνονται τα λεφτά των φορολογουμένων. Τι μπορεί να κάνει γι' αυτό η Επιτροπή. Ο συνάδελφος κύριος ε, Κράμα μίλησε για ανεπαρκείς ε, σιδηροδρομικές διασυνδέσεις με τις χώρες του πρώην παραπετάσματος μεταξύ Πράγας και Δρέσδης. Θέλουμε καλύτερη σύνδεση. Μπορεί να γίνει. Αυτό ήθελα να σου πολύ συγκεκριμένα. Thank you, ε, κυρία Φεραίρα, δύο λεπτά. Έχω δύο ερωτήσει, κύριε Επιτροπέ. Πολλές χώρες έχουν, αντιμετωπίζουν μακροοικονομικά πολύ σοβαρά προβλήματα. Και είναι υποχρεωμένα σε χώρες αυτές που δεν ήταν και από πιο εύπορες να περικόψουν δαπάνε και επενδύσεις. Και στην Πορτογαλία τα μεγαλεπίβολα σιδηροδρομικά προγράμματα δυστυχώς αναθεωρούνται και αναβάλλονται. Κύριε Επίτροπε, έχετε επίγνωση αυτή τη διαδικασία. συνεργάζεστε με αυτές τι χώρες που αντιμετωπίζουν ε, τεράστια οικονομικά προβλήματα προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε πιο διαρθρωτικές επενδύσεις και να μην χαθεί αυτή η δυναμική της σύγκλησης. Δεύτερη ερώτηση για τη βοήθεια, την ενίσχυση προς τις αεροπορικές εταιρείες. Τι θα γίνει με τις χώρες που εξαιτία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν ε, δίνανται να χρηματοδοτήσουν τις αεροπορικές εταιρείες για να αντισταθμίσουν ε, τις απώλειές τους από το νέφος Βεστιακή Ευχαριστώ. Και εγώ έχω μια σύντομη ερώτηση κύριε Επιτροπέ που απορρέει από αυτά που είπε η κυρία Φερέρα για την αντιστάθμιση, την αποζημίωση, δεν ξέρω πώς θα την χαρακτηρίσετε, ή την κρατική ενίσχυση προς αεροπορικές εταιρείες που ζημιώθηκαν από τη διακοπή των πτήσεων εξαιτία του νέφους ηφαιστιακής τέφρας. Κατά τη γνώμη μου, η κατάσταση της κάθε εταιρεία θα εξαρτηθεί από τη γενεοδορία που θα δείξει η χώρα στην οποία βρίσκεται. Ορισμένε χώρες είναι πολύ πιο γενναιόδορες στις κρατικέ του ενισχύσει από ό,τι άλλε. Πιστεύω λοιπόν ότι οποιοδήποτε ε, αεροπλάνο έχει καταχωρηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβει αποζημίωση και εκεί έγκυται η αδυναμία του συστήματος στη διαφορά της δυνατότητας κρατικών ενισχύσεων. Εμείς έχουμε ένα ε, σύστημα ενισχύσεων που δυστυχώς δεν στηρίζεται στον θεμητό ανταγωνισμό. Και γι' αυτό η Επιτροπή μας επέμεινε ότι μέτρο υιοθετηθεί να έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα και να μην παθαθεί στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Κύριε Επίτροπε, ακούμε τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις Ίσως δεν κατάλαβα όλες τις λεπτομέρειες των ερωτήσεων και όλες τις λεπτές τους πτυχές. Μπορείτε να τις ξαναθέσετε. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, είναι ένα θέμα που αναφέρθηκε από πολλούς και έχω την αίσθηση ότι η χρηματοδότηση όντως είναι δύσκολο θέμα και οι προπολογισμοί είναι περιορισμένοι, αλλά οι επενδύσεις στις υποδομές μπορούν να δώσουν όθηση και στην ίδια την οικονομική ανάπτυξη. Βέβαια υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί και υπάρχει δημοσιονομική λιτότητα αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα σε Σαραγώσα. Θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τον, τη χρηματοδότηση από ιδιωτικού φορεί, από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τα περιφερειακά κονδύλια, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από διάφορε πηγέ. Αλλά σήμερα δεν μπορώ να σα δώσω μια ικανοποιητική απάντηση. Δεν έχω κανένα κρυμμένο κορβανά για να χρηματοδοτήσω τα διευρωπαϊκά δικτύα μεταφορών. Θα πρέπει να βρούμε πηγές χρηματοδότησης. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή σα ήταν πολύ σημαντική. Αυτή ήταν βασική ανησυχία και των αεροπορικών εταιριών. Αν δοθούν ενισχύσεις, ε, να εφαρμόζονται με ίσο τρόπο. Μέχρι στιγμής όμως δεν ακούσαμε κανένα παράπονο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει οποιοδήποτε αίτηση για κρατική ενίσχυση με πολύ κριτικό πνεύμα. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβληθεί τέτοια αιτήματα για κρατική ενίσχυση και εμείς πιστεύουμε ότι σε καμία περίπτωση κρατική ενίσχυση δεν θα πρέπει να δημιουργήσει αθέμητο ανταγωνισμό ή στρέβλωση ανταγωνισμού μεταξύ των αεροπορικών εταιριών. Σε ό,τι αφορά τη, τους ερασιτέχνες πιλότους, τι να σας πω, δεν ξέρω τι να πω. Είμαι απροετοίμαστο. Σας υπόσχομαι όμως ότι θα το διερευνήσω και θα σας στείλω πιο τεκμηριωμένη απάντηση για τις αεραστεχνικές πτήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, παρακολούθηση στην ε, Βόρεια και Βαλτική θάλασσα. Δεν ξέρω σε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφέρεστε. Άγια φιάφη. Ναι, όντως, το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προτιμώ να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή πιο διεξοδικά, γιατί όντως υπάρχει πρόβλημα. Υπήρξε ομόφωνη αποδοχή των κρατών μελών που συμμετέχουν στη διεθνή, στο Διεθνή Θαλάσσιο Οργανισμό για να θεσπιστούν κάποια κατόφλια και για θείο και για άλλες ουσίες. Και τώρα ξαφνικά όλοι αρχίζουν και βλέπουν πόσο περίπλοκο είναι το θέμα. Ποιος θα καταρτήσει αυτή τη μελέτη επιπτώσεων. Και το λέω αυτό και στις επιχειρήσεις. Μπορούμε τώρα ξαφνικά να αλλάξουμε τη στάση μας για το θιάφι και άλλες ε, χημικές ουσίες και να ζητήσουμε περιορισμό κάποιων αερίων. Είναι πολύ δύσκολο να ζητήσουμε εξαίρεση ή αναβολή. Προς το παρόν θα έλεγα ότι δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο και μην είμαστε ουτοπιστές. Θα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και ρεαλιστές. Η απόφαση είναι ήδη λυμένη και τα συμπεριφορημένα πρέπει να τηρηθούν. Όταν αποφασίζουμε κάτι πρέπει να το εφαρμόζουμε κιόλα. Γιατί τη στιγμή που λαμβάνεται μια απόφαση μπαίνει σε κίνηση η διαδικασία εφαρμογή τη. Δεν μπορούμε να επαναχωρούμε λοιπόν. Πάντω το θέμα μπορεί να είναι κάπω τεχνικό, αλλά πολιτικά δεν έχουμε μεγάλο περιθώριο ελιγμών. Τώρα, χρονοβόρε ε, εκδόσει δικαστικών αποφάσεων η κατάρτιση ναυτικών τρίτων χωρών, σημαντικό τμήμα του πακέτου για την αυσιπλοεία. Στην Ασία, για παράδειγμα, η κατάρτιση των ναυτικών είναι επαρκής. Υπάρχει σωστή αντιμετώπιση και αξιόλογη κατάρτιση αλλά δεν ξέρω αν ο Διεθνής Οργανισμός για την Αυσιπλοεία ασχολείται και με τα προγράμματα κατάρτισης ναυτικών. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του σιδηροδρομικού πακέτου, είναι ένα θέμα που το έχουμε εξετάσει πολλές φορές. Έχουμε κινήσει ήδη 31 διαδικασίες επί παραβάση κατά χωρών μελών και 21, συγγνώμη, 21 διαδικασίες επί παραβάση και ελπίζουμε να βελτιωθεί ο βαθμός εφαρμογής του σιδηροδρομικού πακέτου από τα κράτη-μέλη και να διαρευνήσουμε με επικοδομητικό πνεύμα όλες τις πιθανές λύσεις. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τα λιμάνια, είναι τμήμα τη ε, στρατηγική μα για την αυσιπλοεία. Τι επαναφορά τη οδηγία για τα λιμάνια εννοείται. Εγώ είμαι υπέρ της απελευθέρωσης των λιμενικών υπηρεσιών. Αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο και δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό είναι τμήμα της ε, στρατηγικής μας, της για την αυσιπλοεία. Θα δούμε πώς θα το χειριστούμε αργότερα. Πάντως, μερικά εμπόδια που υπάρχουν και κολλήματα πραγματικά είναι γελία στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε λοιπόν που απαντήσατε στις ερωτήσεις που ετέθησαν. Ίσως να μην, σας, να μην μας άρεσαν οι ερωτήσεις ή οι απαντήσεις αλλά τουλάχιστον δώσατε κάποιες απαντήσεις. Κοιτάξτε, εμείς ε, προσβλέπουμε στο να συνεχίσουμε το διάλογο μαζί σας ε, σε τακτά χρονικά διαστήματα και τα καταφέραμε να μην καθυστερήσουμε γιατί ξέρουμε ότι είσαστε πολύ επασχολημένος. Σας ευχαριστούμε και πάλι και ευχόμαστε να τα ξαναπούμε σύντομα. Και μερικοί από εμάς θα σας